και εξαντλήσαμε αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη. Η επόμενη σύνοδο θα αρχίσει αύριο, 5η, 11 Φεβρουαρίου 2010, από τις 9.